Αν όχι, εγκρίνονται τα πρακτικά. Να κάνω και κάποιες ανακοινώσεις. Η πρώτη αφορά την κυρία Ιζαμπέλα Ντιμαρτίνη, η οποία μου διαβίβασε ότι προσχώρησε στην ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών από τις ομάδες των Σοσιαλιστών και των, ε, του ECR και του Μία Εγγεγραμμένων. Ε,